Πρώτα για την ε, εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο κύριος Μπονσινιόρε. Με την ψήφο αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή το οποίο η εντολή ε, θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της δικής μας θητείας. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η ψήφος αυτή είναι θετική για όλους μας, για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής θα ασχοληθεί ε, με, τα, ε, με, τα παράπονα των πολιτών έναντι της κακοδιοίκησης σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών. Ε, ο διαμεσολαβητή απάντησε σε ερωτήσει του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση τη διαφάνεια, τη εργασία του, τη βελτίωση της συνεργασία ε, των υπηρεσιών του με ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ρόλο του θα είναι πολύ σημαντικό για την προάσπιση των Ευρωπαίων πολιτών, για να του βοηθήσει στη σχέση του με τη δημόσια διοίκηση και ενδεχομένω για να ακουστεί η φωνή των πολιτών και να καταλάβουν οι πολίτε ότι η Ευρώπη αποτελεί ένα σύνολο κοινών θεσμών θεσμών. Για την καταπολέμηση επίση γραφειοκρατία. Στόχο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε όλους, όλοι μα. Θα πρέπει λοιπόν να θέσει το επίκεντρο τη δράση του τον πολίτη. Και εκφράζω την ευχή ε, ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να αξιοποιήσει την εμπειρία του του παρελθόντο για να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι θετικέ του σχέσει με την Ευρώπη των πολιτών. Ευχαριστώ. Στην έκθεση της κυρίας Τζολί έχουμε πέντε αιτιολογήσεις. Πρώτο ο κύριος Αντωνιώτση. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ε, η κυρία Ζολή ε, εργάστηκε με εξαιρετικό τρόπο ε, και συνεργάστηκε ιδιαίτερα με όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, υποστηρίζω ιδιαίτερα θερμά ε, με τους συναδέλφους του ΕΛΚ την έκθεση αυτή. Και θα ήθελα να υποστηρίξω ιδιαίτερα και να εκφράσω την υποστήριξή μου στο τμήμα αυτό της ε, έκθεσης όπου υπογραμμίζεται το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της συμφωνίας ε, της, του Κοτονού θα πρέπει να λάβουν υπόψη από τη μια τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και από την άλλη τα φαινόμενα μετανάστευσης κυρίως ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη ε, αντιμετώπισης και αναχέτησης παράνομης μετανάστευσης. Διότι ε, είναι ιδιαίτερα αρνητικός ο αντίκτυπος του φαινομένου αυτού τόσο στις οικονομίες των χωρών ΑΚΕ, διότι λόγω αυτού του φαινομένου χάνουν εργατικό δυναμικό και μάλιστα εργατικό δυναμικό ιδιαίτερα εξειδικευμένο που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη, αλλά κατά ταυτόχρονα όλα αυτά είναι εις βάρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως αυτών που πλήττονται ιδιαίτερα από την παράνομη μετανάστευση. Όπως η Ιταλία που πλέον ε, δεν έχει ικανότητα απορρόφηση των μεταναστών αυτών. Από άποψη απασχόληση, από οικονομική άποψη έχουμε φτάσει στα όρια μας και ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα κοινωνικού εκφυλισμού. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα κατά της έκθεσης Ζολή αν και συμφωνούμε όλοι για τις βασικές αξίες, ότι θα πρέπει να ασκήσουμε μια πολιτική για την προώθηση, την ανάπτυξη των αφρικανικών χωρών, προκειμένου και οι Αφρικανοί να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην ε, εξέλιξη και την πρόοδο της χώρας τους. Το καταλαβαίνω αυτό και το υποστηρίζω. Γιατί όμως στην ίδια έκθεση τεσόμαστε τόσο πολύ υπέρ μιας νέας ε, μετανάστευσης από τις αφρικανικές χώρες, για μια μετανάστευση προς την Ευρώπη. Αυτό ε, προωθεί το brain drain, τη διαφυγή εγκεφάλων των πιο ικανών Αφρικανών. Και αυτή η μπλε χάρτα που είναι πολύ ε, λαβερή και για την Αφρική αλλά και για την Ευρώπη. Και αυτή η εκπεριτροπή μετανάστευση είναι κάτι το πολύ αμφιλεγόμενο, γιατί δεν επιστρέφουν ποτέ οι μετανάστες και δημιουργούν νέους παράνομους μετανάστευση. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ατζέντα μας ήταν αρκετά ε, ασθενείς αυτή την εβδομάδα. Γιατί, γιατί υπήρξαν ελιγμοί, αλλά στις Βρυξέλλες. Και περάσαμε σε ακροάσεις και τώρα καλούμαστε να ορίσουμε τους 27 καλύτερους ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα είναι μόνο το εκτελεστικό σώμα, αλλά θα έχουν και δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας υποβολή ε, προτάσεων. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη γιατί δεν είναι άμεσα υπόλογοι στο, στο εκλογικό σώμα. Και αυτό κλήθηκαν να αποφασίσουν όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ευρωσκεπτικιστής για να το βρίσκει αυτό παράλογο. Μου φαίνεται περίεργο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε μια διαδικασία τόσο ταπεινωτική για όλους μας. Ο κύριος Καμάλ για ένα λεπτό. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξετάζοντας τις σχέσεις μεταξύ και, και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη αρχή θα πρέπει να είναι πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο να εξέλθει από το καθεστώς στόχιας. Και πολύ συχνά ο κόσμος στις χώρες αυτές παραπονιούνται γιατί 40 χρόνια μετά την ανεξαρτησία τους ακόμα υποφέρουν από τα, 40, από τα χρόνια του σοσιαλισμού που εξαρτώνται από τις πρωτεύουσες οικονομίες και οι επιχειρηματίες στις χώρες αυτές μου λένε ότι τα, οι εμπορικοί φραγμοί κάνουν δύσκολε και πιο ακριβές τις εισαγωγές τροφίμων για τους πιο φτωχούς πολίτες ε, παραπονιούνται για τους δασμολογικούς και μη φραγμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση σύστησε μία ομάδα για να ενισχύσει τους επιχειρηματίες ε, των χωρών αυτών για να εξάγουν στην Ευρώπη. Και ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη αρχή είναι να προωθήσουμε τους επιχειρηματίες στις φτωχές αυτές χώρες και το εμπόριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και μόνο η παράγραφος 31 της έκθεσης της Ευαζολής ήταν αρκετή για να μας κάνει να τις καταψηφίσουμε, όπου καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει την αρχή της περιστροφικής ε, ε, μετανάστευσης και των σχετικών θεωρήσεων. Αυτή η μετανάστευση είναι μια φάτα μουρκάνα, γιατί υπάρχουν επίσημα έγγραφα Υπάρχει μόνο στα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι στην πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό, ότι ένας μετανάστης ε, λαμβάνει μια άδεια παραμονής περιορισμένης διάρκειας, αλλά παραμένει μετά την ε, λήξη της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως λάθρο μετανάστης. Αυτή είναι η πραγματικότητα της μετανάστευσης αυτής. Αποτελεί, αν θέλετε, μία άλλη λέξη για την λάθρο μετανάστευση. Το ξέρει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά το προωθεί γιατί ο κόσμος ε, θεωρεί ότι πολλοί μετανάστευση επιστρέφουν στη χώρα προέλευσή τους. Θα ήταν ε, λοιπόν καλό να σταματήσουμε να καμουφλάρουμε με τέτοιο τρόπο την πραγματικότητα. Και τέλος ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την άδειά σα θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά ε, το χρονοδιάγραμμα και την τήρηση του χρόνου. Γιατί πάρα πολύ συχνά εδώ ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πάρα πολύ ξεπερνούν το χρόνο του και του επιτρέπεται. Ορισμένοι διπλασιάζουν το χρόνο που έχουν στη διάθεσή του. Απευθύνω έκκληση στου διάφορους προεδρεύοντε να χρησιμοποιήσουν την αρμοδιότητά του, έτσι ώστε να τηρούν το χρόνο σύμφωνα με του κανόνε. Και επίσης ε, όσον αφορά την διαδικασία κάτι θα πρέπει όλοι να έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε. Ευχαριστώ. Λίγη συνεδρίαση και αρχίζει εκ νέου στι 3 ώρα το απόγευμα.